Καλημέρα σα, κύριε και κύριοι. Το Της είναι η δήλωση για την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμφουλίου. Το λόγο θα πρέπει να πάρει ο κύριος Φαν αλλά απουσιάζει. Άρα πρέπει να τον περιμένουμε.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 και εγώ μπορώ να σας διηγηθώ διάφορα για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, άμα θέλετε να ακούσετε τα δικά μου σχόλια, αλλά... Α, ωραία, ωραία, ωραία. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Είχαμε ξεκινήσει τη συνεδρίαση και έχετε το λόγο, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1η και 2η Μαρτίου ήταν